Άρχεται η σημερινή συνεδρίαση, έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιπολογισμών. Θέλω να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω την κυρία Γεωργίευα για την παρουσία της. Μόλις έφυγε από συνεδρίαση του Σώματος των Επιτρόπων και έρχεται να ενημερώσει αμιλητή την Επιτροπή Προϋπολογισμών για το περιεχόμενο του διορθωτικού προϋπολογισμού 2015 υπαριθμούν 7. Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 7 αφορά το μεταναστευτικό και το προσφυγικό και τι λύσεις μπορούν να δοθούν στις ε, χώρες που υποδέχονται το μεγάλο αυτό αριθμό ατόμων. Η αρμόδια λοιπόν επίτροπος ε, θα προτείνει κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για τις ε, αναλήψεις αυτές υποχρεώσεων, για αυτές τις δεσμεύσεις που είναι πάνω από την οροφή. Φαντάζομαι ότι αυτό θα σημαίνει κάποιες ε, ελαφρύσεις στις ε, πληρωμές. Να δούμε αν και αυτές θα είναι πάνω από το όριο, το ανώτατο ή όχι. Ε, θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω για τις ε, Αποφάσει που ελήφθησαν στην χθεσινή συνεδρίαση των συντονιστών. Αποφασίσαμε να διοργανώσουμε τρει δημόσιε ακρόασει ενώπιν τη Επιτροπή Προπολογισμών και αυτό θα γίνει στο πρώτο εξάμεινο του 2016. Η Πρώτη ακρόαση θα αφορά την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Η ημερομηνία θα ειναι ιανουαριο Ιανουάριο-φεβρουάριο. Δεύτερη ακρόαση με θέμα τα νέα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία και το ρόλο των National Promotional Banks υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κατά το Μάρτιο τη βλέπουμε αυτή την ακρόαση. Και τέλος, τρίτη ακρόαση για τις μεσονομικές επιπτώσεις της ε, κρίσης ε, που έχουμε σήμερα με τους πρόσφυγες, τους ετούντες άσυλο και τους μετανάστες, η οποία ακρόαση θα γίνει σε συνεργασία με άλλες στις αρμόδιες ενδιαφέρομενες επιτροπές, ε, τη ΛΥΜΠΕ συγκεκριμένα, για την εσωτερική εξωτερική διάσταση του προβλήματος αυτού και κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει το Μάιο η ακρόαση αυτή. Επίσης οι συντονιστές αποφάσισαν ότι εγκρίνονται τέσσερις ε, αποστολές, ε, διαπροσωπιών η πρώτη το Φεβρουάριο στην Τουρκία, στην Πράσινη Εβδομάδα, η δεύτερη σε Λίβανο, η Ορδανία το Μάη, γιατί είμαστε σε επικοινωνία και αυτό έχει να κάνει και με όσα θα μας πει Επίτροπος. Τρίτη αντιπροσωπεία Βερολίνο-Παρίσι για να γίνει απολογισμός της δημοσιονομικής κατάστασης και των συστάσεων. Μεταξύ Μαρτίου-Απριλίου θα γίνει αυτή και η τέταρτη τον Ιούλιο στην Ελλάδα. Τέταρτη αποστολή για να δούμε επιτόπου και με βάση αποδεκτικά στοιχεία όσο αποδίδουν τα μέτρα των δημοσιονομικών, των, τα δημοσιονομικά μέτρα και τα διαρθρωτικά μέτρα που έχουν υιοθετήσει οι ελληνικές τοπικές αρχές. Αυτά λοιπόν, να σας πω επίσης ότι λάβατε με ηλεκτρονικό ταχυδρομή στις 11 τις αδρές γραμμές της πρότασης για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας αλλά θα μας τα πει και η κυρία Γεωργίευα. Κυρία Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που δεχθήκατε να έρθετε και να μας ενημερώσετε σε πραγματικό χρόνο στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Σας δίνω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε να παραστώ ενώπιον σας σήμερα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Προπολογισμών. Όντως το Κολέγιο Επιτρόπων μόλις ενέκρινε τον διορθωτικό προϋπολισμό 7-2015 ως τμήμα της συνολικής μας ανταπόκρισης στην κρίση του προσφυγικού. Προβλέπει σημαντική αύξηση χρηματοδότησης. Διπλασιάσαμε συνολικά τα χρήματα που διαθέτουμε για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Από 4,5 δισεκατομμύρια στις αρχές του έτους φτάνουμε στα 9,2 δισεκατομμύρια. Όχι μόνο δηλαδή αυξάνουμε σημαντικά τη χρηματοδότηση που προσφέρουμε, αλλά και ελπίζω να έχουμε εκεί την υποστήριξη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών, θα τα κάνουμε αυτά και σε χρόνο ρεκόρ Κατανοείται βεβαίως για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντικό αυτό, δηλαδή να δείξουμε στους Ευρωπαίου πολίτες ότι είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε με ταχύτητα για να ε, ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες τους. Να πω τώρα στις λεπτομέρειες της προτάσεως μας. Όπως είπα προηγουμένως, αρχίσαμε το 2015 με 4,5 δισεκατομμύρια για το 2015-2016. Μετά προτείναμε μέτρα που έφταναν το ύψος των δισεκατομμυρίων, ιδίως για τη χρηματοδότηση του προγράμματος μετεγκατάστασης 160.000 ε, μεταναστών και προσφύγων έτσι ώστε να είναι συνολική η ευρωπαϊκή απάντηση και ένα πρόσθετο πακέτο για το 2015-2016 που ανακοινώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου. Ένα δισεκατομμύριο από αυτό το τελευταίο πακέτο πρόκειται να διατεθεί για εξωτερικές δράσεις, για να ε, συνδράμουμε τους ανθρώπους έτσι ώστε να παραμείνουν εκεί όπου βρίσκονται τώρα, δηλαδή στις γειτονικέ χώρες της Συρίας, καθώς και για κάποιες ανθρωπιστικές δράσεις εντός της Συρίας. 700 εκατομμύρια ευρώ για εσωτερικά μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτηθούν μέτρα που λαμβάνουν οι χώρες μέλη και για να ενισχυθούν οι μεθοριακοί έλεγχοι. Φτάνουμε λοιπόν στα 7,5 δισεκατομμύρια. Εδώ προσθέτουμε 1,8 δισεκατομμύρια για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αφρική, Transfund, που χρηματοδοτούνται κυρίως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αναπτύξεως και να υπενθυμίσω ότι στην διάσκεψη αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων την προηγούμενη εβδομάδα ανέλαβαν την δέσμευση να κινητοποιήσουν ένα πρόσθετο ποσό ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για να ενισχύσουν τον ύπατο αρμοστή των ΕΕ για τους πρόσφυγες καθώς και το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Διατροφών, Διατροφής συγγνώμη, και άλλους σημαντικούς οργανισμούς επιτόπου, που δρούν επιτόπου όπως ACIRC. Πρόσθετο λοιπόν ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Να έλθω τώρα στις δύο αποφάσεις που εγκρίναμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρώτη, διορθωτικός προϋπολογισμός 7 του 2015. Πρόκειται για σημαντικότατο μέρος αυτών, αυτής της δέσμης ταχαίων μέτρων για την αντιμετώπιση αυτής της ανευπροηγουμένου κρίσεως. Το δεύτερο, η δεύτερη απόφαση είναι η κινητοποίηση του αποθεματικού επίγουσας ανάγκης. Να το χρησιμοποιήσουμε δηλαδή για το υπόλοιπο ποσό στο αποθεματικό, που βρίσκεται στο αποθεματικό για φέτος. Στο σύνολό τους, οι δύο αυτές προτάσεις επιτρέπουν την κινητοποίηση 800 περίπου χιλιάδων ε, συγγνώμη, 800 ε, εκατομμυρίων, 800 ευρώ ακόμη φέτος, μέσα στο έτος 2015. Μπορούμε να, δηλαδή να κάνουμε σημαντικά βήματα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Αυτός ο διορθωτικός προϋπολογισμός του 7-2015 προβλέπει ενίσχυση στις πιστώσεις υποχρώσεων για μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης του προσφυγικού. στην ε, κατηγορία 3 και στην κατηγορία 4 για εσωτερικά και εξωτερικά μέτρα. Δηλαδή να προσφέρουμε άμεση βοήθεια στις πλέον θυγόμενες ευρωπαϊκές χώρες μέλη, να ενισχύσουμε τους, οργανισμούς, τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς που δρούν στα σύνορα και να ενισχύσουμε και τρίτες χώρες. Αυτά τα 4,3 λοιπόν, δισεκατομμύρια πηγαίνουν κυρίως για το Ταμείο με τη Μετανάστευση και το Προσφυγικό, ΑΕΣΕΦ, 100 εκατομμύρια επίγουσα βοήθεια για τις πιο θυγόμενες χώρες μέλη για την υποστήριξη προγραμμάτων αντιμετώπισης του προβλήματος των μεταναστών και για τη δημιουργία των hot spot, δηλαδή ταχύτατη αύξηση των ικανοτήτων υποδοχής σε χώρες όπου φτάνουν οι μετανάστες και πρόσφυγες σε μεγάλους αριθμούς. 120 εκατομμύρια ακόμη για τους οργανισμούς, για τους οργανισμούς του, ε, των Ηνωμένων Εθνών. 60 ε, θέσεις για την, ε, για την Frontex, 30 για την Ευρωπόλ και 30 για την ΑΣΟ. 300 εκατομμύρια για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Γειτονικής Σχέσης για να αντιμετωπίσουν προβλήματα που πρόκειται από την κρίση της Συρίας. Το λεγόμενο, το λεγόμενο Ταμείο Ελπίδος για την ενίσχυση των γειτονικών χωρών της Συρίας που υποδέχονται πρόσφυγες. Γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό. Ένας σημαντικός λόγος που οθεί τους πρόσφυγες να έλθουν στην Ευρώπη είναι διότι έχασαν την ελπίδα. Θεωρούν ότι ο κόσμος τους ξέχασε. Ότι ο πόλεμος ποτέ δεν θα τελειώσει, ότι ποτέ θα επιστρέψουν στις αισθητήρες τους και ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες διαβιούν θα γίνονται όλο και χειρότερε. Αυτό, γι' αυτό λοιπόν λέγεται και το Ταμείο αυτό, το Ταμείο Ελπίδα. Τώρα τα άλλα μέτρα ναι, έχουν ω εξή. 200 εκατομμύρια από το ΑΙΠΑ και ΕΝΗ, λέει η κυρία Γεωργίευα, για να ενισχυθούν το Ταμείο για τη Συρία και να συμπληρωθούν τα 300 εκατομμύρια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Γειτονίας, ΕΝΗ. Άρα θα φτάσουμε πάνω από 500 εκατομμύρια συνολικά για να διατηθούν για την κρίση για τη Συρία. Άλλα 200 εκατομμύρια για ανθρωπιστική βοήθεια. Άμεση ανταπόκρισή μας δηλαδή για τους πρόσφυγες. Μέσω των Ενωμένων Εθνών, του World Food Program και του ECIRC μέσω της έκτακτης ενίσχυσης 10 εκατομμύρια από το αποθεματικό για την ανθρωπιστική βοήθεια, επίση επίσης άλλο από την μεταφορά πιστώσεως που είχε ήδη εγκριθεί και άλλη αίτηση μεταφοράς για 175 εκατομμύρια από το αποθεματικό έκτακτης ανάγκης. Και αυτά είναι που σας έχω δώσει σήμερα. Για αυτές λοιπόν τις άμεσες ενέργειες χρειαζόμαστε πιστώσεις πληρωμών που να φτάνουν το 40% των δεσμεύσεων που έχουμε ήδη αναλάβει, δηλαδή πιστώσεις πληρωμών της τάξης των 70 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο διορθωτικό προϋπολογισμό 7. Εκεί να περιληφθούν και 30 εκατομμύρια από το Emergency Aid Reserve και τα υπόλοιπα θα πάνε για το 2016. Παρά αυτόν τον διορθωτικό προϋπολογισμό 7-15, και τα πράγματα που εγκρίναμε στην Κομισιόν, αυτά σας παρουσιάζω τώρα, δώσαμε και τη λεγόμενη Global Transfer για να ολοκληρωθούν προγράμματα για την ασφάλεια των συνόρων, για την ασφάλεια και την αντιμετώπιση κρίσεων, δηλαδή κατηγορίες 3 και 4. Και τα υπόλοιπα πηγαίνουν κυρίως για να πληρωθούν οι ανάγκες προγραμμάτων προγραμμάτων όπως ο Έρασμος, εκεί πηγαίνουν 170 εκατομμύρια. Εγώ θα ήθελα να απευθυνθώ σε σας και να ζητήσω την υποστήριξή σας. Χρειαζόμαστε ταχεία έγκριση της συνολικής δέσμης που περιλαμβάνεται στο διορθωτικο προϋπολογισμό προϋπορισμό 7-2015, το Emergency Aid Reserve και το Global Transfer για να μπορέσουμε να διαθέσουμε λοιπόν τις πιστώσεις αυτές το δυνατόν συντομότερο και ιδίως για την έξτρα χρηματοδότηση για το παγκόσμιο πρόγραμμα διατροφής διότι λείπουν τα τρόφιμα σε πολλά στρατόπεδα προσφύγων και στο Λίβανο και στην Ιορδανία γι' αυτό έχει τεράστια σημασία να δοθεί το μήνυμα ότι έρχεται η ευρωπαϊκή βοήθεια φτάνει βλέπω να εκπροσωπείται και το Συμβούλιο. Την ίδια έκκληση απευθύνουμε και στο Συμβούλιο. Παρακαλούμε να εγκρίνετε ταχύτατα τα εν λόγω μέτρα. Δυστυχώς, με τα μέτρα που λαμβάνουμε, δεν πρόκειται βεβαίως να αποσοβηθεί η κρίση. Θα χρειαστεί λοιπόν να εξετάσουμε και τον προϋπολογισμό του 2016 έτσι ώστε να γίνει και αυτός ένα ισχυρό εργαλείο στην ανταπόκριση που έχουμε για την κρίση. Μέσα Οκτωβρίου θα αποστείλουμε επιστολή για, να, για τις αποφάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης και στην φετινή διαδικασία του προϋπολογισμού θα έχει πολύ μεγάλη σημασία Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δείξουν ότι εμείς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούμε να συνεργαστούμε και να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας βεβαίως μέσα στην περίοδο διαδικασίας συνδιαλλαγής. Κύριε Πρόεδρε και εσείς αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, πιστεύω ότι η παρουσίαση που σας κάνω δείχνει πόσο σοβαρά λαμβάνουμε υπόψη την κρίση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου εδώ της Γενικής Διευθύνσεως Προϋπολογισμών, αλλά και βεβαίως και σε όλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εργάζονται νυχθημερών και δεν φύρονται καμιάς προσπάθειας για να βρούμε τα απαραίτητα κονδύλια και να τα θέσουμε υπό την έγκρισή σας. Ασφαλώς πρόκειται για την υψηλότατη προτεραιότητα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και δεν έχω αμφιβολία ότι θα ανταποκριθούμε στην πρόκληση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Αντιπρόεδρε για δώσουμε μας ανακοινώσατε. Δευτέρα και Τρίτη πρόκειται να συνεδριάσουμε και θα συζητήσουμε το σύνολο των ε, τροπολογιών και των ε, ε, συμβαστικών που ο Γενικό Συγητή μπόρεσε να σύγκεντρώσει με τη σύμφωνη γνώμη όλων των πολιτικών ομάδων και να θυμηθούμε ότι πριν από μια εβδομάδα οργανώσατε αυτό το αξιόλογο φόρουμ που αφορά τον προπολογισμό για να διαπιστωθεί πόσο χρειάζεται η ευελιξία και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το 2015 είναι πλήρες ε, γεγονόντων που μας ε, οθούν τόσο ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε περισσότερη ευελιξία σε αυτό το άκαμπτο πλαίσιο. Είπαμε ότι έχουμε ορθοτικές κινήσεις για τον προηγουσμό της Γεωργίας, είπαμε και αυτά τα 500 εκατομμύρια αλλά η διορθωτική πρόταση θα αφορά και τον προπολογισμό της χρήσης του 16 όσον αφορά την ενίσχυση για τους ε, πρόσφυγες και τις χώρες που τους αναδέχονται και αυτό να γίνει όσο γίνεται πιο σύντομα. Μην μετοπιστεί δηλαδή αυτή η κρίση που δυστυχώς θα πάει πέρα από το 15 και το 16. Και προβληματιζόμαστε γιατί βλέπουμε το πόσο δύσκολη δουλειά έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστούμε να τώρα τον ε, λόγο στην Γενική Συγκίτρια για το 2015, κύριε Γαρτιά Θάμπορ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε που ήρθατε τόσο γρήγορα για να μας παρουσιάσετε τον διορθωτικό προπολογισμό και ε, εγώ παίρνω όλα αυτά τα έγγραφα, προσπαθώ να δω την ε, πρότασή σας στις λεπτομέρειές της και ε, όπως είπαμε ενεργούμε όσο γίνεται ταχύτερα και όπως είπατε και εσείς πρόκειται για την ύψιστή μας σημερινή προτεραιότητα για να υπάρχουν αρκετοί και διαθέσιμοι πόροι ούτως ώστε να ανασχέσουμε την κρίση με τους πρόσφυγες να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας από πλευράς προϋπολογισμού. Και όπως λέγατε, με ακούτε, λειτουργεί η μετάφραση. No problema. Decía que, Σας έλεγα ότι σας ευχαριστούμε που ήρθατε τόσο γρήγορα. Αντιδράσετε για να παρουσιάσετε την πρόταση για διόρθωση του προϋπολογισμού. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές και εμείς ε, σαν Κοινοβούλιο ε, είναι θέμα προτεραιότητας να ανασχέσουμε την κρίση με το μεταναστευτικό με τους απαραίτητους πόρους. Δεν έχουμε ακόμα μελετήσει τις λεπτομέρειες της πρότασής σας, αλλά ε, σίγουρα και θα ασχοληθούμε όλοι μας και θα προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα για να εγκριθεί το συντομότερο διορθωτικός προπολογισμό για να εκταμιευτούν αυτά τα κονδύλια. Ξέρω ότι τα περισσότερα τα γράφετε στα έγγραφα, αλλά τι γίνεται με αυτά τα 70 εκατομμύρια τα οποία θα ξαναδιαθέσετε. Για πέστε μου ποια, ποιες γραμμές, ποια κονδύλια θα καλυφθούν, γιατί υπάρχουν τα χρήματα τώρα και εσείς ε, θέλετε να τα ξαναεντάξετε στον προηγούμενο του 16. Τώρα όσον αφορά τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, όπως γνωρίζετε, υπάρχει κάποια προστριβή όσον αφορά το προσωπικό αυτόν, ΕΑΣΟ, Europol και Frontex και για πέστε μου στη διορθωτική πρόταση για το 16 τι θα κάνετε θα αφήσετε αμετάβλητο το προσωπικό αυτών των υπηρεσιών και επίσης έχω ένα δισταγμένο φόβο για το μέλλον όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών για άλλη μια φορά γιατί είδαμε τι, τι, τι, τι πρόταση υπάρχει για την Ελλάδα, δεν υπάρχει αλλαγή, κρίθηκαν αλλαγή και τώρα υπάρχει αυτή η πρόταση αύξησης της πληκοδότησης που δεν θα έχει συνολικά ε, συνέπειες στις πιστός πληρωμών, αλλά τι γίνεται, μήπως ε, με αυτή την αύξηση μπορέσουμε κάτι να κάνουμε με τα, όλα αυτά τα ανεξόφλητα που υπάρχουν, γιατί το 16 Πρέπει να πετύχουμε αυτό το στόχο, αλλά τα χρήματα από κάπου θα βγουν για να διατεθούν. Άρα πετύχουμε το στίχο στο 16, αλλά μήπως έτσι υπονομεύσουμε τους άλλους στόχους του απότερου μέλλοντος. Οπότε θα πρέπει να ξανατσεκάρουμε τους λογαριασμούς μας και να δούμε τι θα γίνει στα πλαίσια ε, των διευθυντικών προοπτικών. Και βεβαίως από την αρχή η Κομισιόν πήρε στα σοβαρά το θέμα της μεταναστευτικής κρίσης. Εμείς εδώ είμαστε. Οπωσδήποτε θα σας βοηθήσουμε. Και θα πρέπει όλοι, αλλά και το Συμβούλιο, να είμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Ο Πρόεδρος. Και τώρα, οι συντονιστές. Φερνάντες. Σας ευχαριστώ. Παίρνω το λόγο και ως συντονιστής και ως εισηγητής για το προϋπολογισμό του 2016. Θέλω να καλωσορίσω την Επιτρόπου και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να την ευχαριστήσω για την ε, προθυμία που επέδειξε, τη διαθεσιμότητά της, όπως πάντοτε άλλωστε ε, είναι διαθέσιμη να μας συναντά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία ε, Γεωργίευα που ήρθατε εδώ να μας ε, παρουσιάσετε άμεσα τον διορθωτικό προπολισμό 7 που ουσιαστικά τα σε μια επίγουσα ανάγκη. Εμείς είχαμε αναφέρει και τον Ιούλιο το ζήτημα της κρίσης, το προσφυγικό ζήτημα, το είχαμε χαρακτηρίσει κατεπήγον θα πρέπει λοιπόν να, ε, ε, τα λόγια μας ε, να συνάδουν με τα έργα μας. Είπαμε ότι η αλληλεγγύη είναι κάτι που δεν μένει στα λόγια, αλλά πρέπει να γίνεται πράξη. Πρέπει να είμαστε συνεπείς και θέλω να πω ότι με ικανοποιεί ακριβώς γι' αυτό το λόγο ιδιαίτερα η πρόταση ε, και η διάσταση που δίνεται για την επίλυση του ζητήματος ε, στο εσωτερικό, έχουμε την κατηγορία 3, αλλά και την εξωτερική διάσταση καλύπτουμε. Έχουμε λοιπόν μια δέσμη μέτρων για την επίλυση του σημαντικού αυτού ε, προβλήματος. Θα πρέπει να έχουμε συνδυασμό κατηγορίας 3 και 4, το αποθεματικό έμπλεξης βοήθειας και όλα τα άλλα μέσα για την ανάπτυξη, για τη συνεργασία οργανισμοί, όπως ε, έχω προείπει άλλωστε εδώ, ε, θεωρώ ότι είναι απαραδεκτό το Συμβούλιο για την κατηγορία 4 να προτείνει περικοπές σε μέσα και μηχανισμούς που θα μπορούσαν να περιορίζουν ε, τέτοια προβλήματα. Πρόκειται για μια έκτακτη κατεπίγουσα περίσταση Πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υπάρχει συμπληρωματική βοήθεια, συμπληρωματικός προπολογισμό. Εδώ λοιπόν τώρα δείχνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε, όπως είπα, μια κατεπίγουσα ε, περίσταση που απαιτεί συμπληρωματικούς πόρους. Χαίρομαι λοιπόν που θα χρησιμοποιήσουμε το μηχανισμό ευελιξίας, το αποθεματικό επίδουσας βοήθειας. Αλλά θέλω να μου διευκρινίσετε δύο πράγματα. Το 2015 συγκεκριμένα ποιο είναι το συμπληρωματικό ποσό που δεν είναι ε, απόρρια ανά διανομής κάποιων πόρων. Ποιο είναι δηλαδή το έξτρα ποσό που προτείνεται για το 2015. Επίσης, θέλω να μου πείτε για το 2016 ποιος θα είναι ο αντίκτυπος της κατάστασης για τη συγκεκριμένη αυτής πρότασης της ε, ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παραλαμβάνω ποιος θα είναι ο αντίκτυπος για το 2016. Αν μπορείτε να προκαταλάβετε ήδη κάπως τα πράγματα. Διορθωτικός Οκτωβρίου 2016 εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός με πολύ μεγάλη πλειοψηφία στην Επιτροπή μας. Αυτή άλλωστε ήταν η εντολή που λάβαμε στο πλαίσιο του τριμέρους διαλόγου. Εδώ μιλώ λοιπόν για μια πολύ αποφασιστική πρόταση που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το μηχανισμό ευελιξίας στην κατηγορία 4. Είμαστε πολύ μετριοπαθείς εφόσον παραμένουμε εντός των περιθωρίων, εντός των όριων. Άρα θέλουμε να ε, παραμείνουμε σε μια λογική λιτότητα από ό,τι φαίνεται. Σε ό,τι αφορά όμως το μηχανισμό ευελιξίας, νομίζω ότι εδώ πρέπει ε, να κάνουμε τη βέλτιστη δυνατή χρήση. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε συνένεση και να κατανοήσουμε όλοι ότι όταν μιλάμε για ένα μηχανισμό ευελιξία, μιλάμε για μέσα που πρέπει να υπερβούν τις οροφές του υπολογισμού. Εκτός οροφής λοιπόν, πάνω από τα ανώτατα όρια που προβλέπονται. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για ευελιξία και μηχανισμό ευελιξίας. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, θέση αυτή την οποία θέτησε. Επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται κατεπίγουσα δράση γιατί μιλάμε για την ανθρώπινη εξωπρέπεια, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, έρχεται χειμώνα. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδιάφοροι. Πρέπει να είμαστε συνεπείς. Είναι καιρός να δράσουμε. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος, Κύριος Κουσμίουκ, εκ μέρους του ECR. Δεν θέλετε το λόγο. Ο κύριος Ντεπχέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με ικανοποίηση σημειώνω ότι φαίνεται να συμφωνεί και ο συνάδελφος με τις προτάσεις της Κομισιόν και χαίρομαι. Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό κυρία. Ναι, η σιγή σημαίνει συνδένεση, συγκατάθεση. Έτσι φαίνεται, μάλιστα. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ που ήρθατε τόσο γρήγορα μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής που ενέκρινε τις προτάσεις τις οποίες μας κοινοποιήσατε. Είναι μια κίνηση την οποία εκτιμούμε, μια χειρονομία την οποία εκτιμούμε ιδιαίτερως. Συνολικά πρέπει να σας πω ότι δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσετε δυσκολία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Επιτροπή μας, αν θέλετε πρώτον να προχωρήσουμε γρήγορα και δεύτερον, ε, αν θέλετε να αξιοποιήσουμε ε, τις προτάσεις σας και να καλύψουμε αυτές τις συμπληρωματικές ανάγκες που κρίνεται αναγκαίες και μας παρουσιάσατε. ...9,6 είναι νομίζω συνολικά τελικά αυτό το ποσό. Ε, για αυτό το ποσό, το συνολικό των 9,6 δις, πολλά θα εξαρτηθούν από τη στάση του ε, Συμβουλίου και από τη συμμετοχή των κρατών μελών για την τροφοδότηση των διαφόρων ταμείων, trust fund για την Αφρική κτλ. κτλ. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή διαβουλεύεστε με τα κράτη-μέλη για να επιδείξουν την ίδια προσήλωση και αφοσίωση ε, όπως αυτή που στείλεται και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θέλω και δεν μπορώ και να επισέλθω στις λεπτομέρειες προτάσεις σας προς το παρόν τουλάχιστον. Άλλωστε δεν έχω μελετήσει ανδελεχώς αυτές τις προτάσεις, αλλά θα ήθελα να κάνω κάποιες σκέψεις. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση του ΑΜΥΦ. δεν ξέρω αν μπορείτε να μου απαντήσετε, οι υπηρεσίες σας τα μπορούσαν. Ο κανονισμός προβλέπει ε, τη διάθεση των κονδυλίων αυτού του ταμείου. Έχω τον ε, κανονισμό, τέλος πάντων δεν θα σας τον διαβάσω τώρα, απλά ήθελα να ξέρω ότι συνάδει ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να διατεθούν τα κονδύλια με τον ίδιο τον κανονισμό γιατί τελείως θα πρέπει να τον τροποποιήσουμε διότι δίνονται συγκεκριμένα κονδύλια σε αυτόν τον κανονισμό, συγκεκριμένες ε, διατάξεις ισχύουν. Θα ήθελα λοιπόν να μου δώσετε τώρα, αν δεν μπορείτε τώρα έστω κάποια άλλη στιγμή, ε, συγκεκριμένα το πώς θα προχωρήσετε. Επίσης, θα χρειαστούν φαντάζομαι νομοθετικές προσαρμογές, γιατί προτείνεται σημαντική ενίσχυση των μέσων ε, του Frontex. Θα έχει και νέα αποστολή Frontex. Θα έχει δηλαδή δικαίωμα πρωτοβουλίας για την οργάνωση επιστροφών, κάτι που δεν έχει αυτή τη στιγμή. Θα χρειαστούν λοιπόν κάποιες επαναλαμβάνω μυθικές προσαρμογές δεδομένης της ενίσχυσης και σημαντικής ενίσχυσης των μέσων που μας αναφέρατε. Δεν το, δεν το συζητήσαμε και δεν έχω μελετήσει κι εγώ αλλά δεδομένου του κατεπήγοντος και των προτάσεων που διατυπώνεται. Τι θα γίνει με τις πληρωμές, ε, όπως τις εκτιμούσατε για το 2016, παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Κάνατε κάποιες εκτιμήσεις. Γιατί ξέρετε ότι εμάς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Και θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να τηρεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει σε αφορά τις πληρωμών για να μην έχουμε αυτά που είχαμε σε προηγούμενες χρονιές. Θα ήθελα κάποια διευκρίνηση πάνω και σε αυτό. Έχω και άλλες ερωτήσεις, αλλά φαντάζομαι θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε όταν θα έχουμε μελετήσει πιο αναλυτικά τις προτάσεις σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαραγκάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος και εν μέρει γιατί θα ήθελα να σας πω ότι συμφωνώ και να μην επαναλάβω αυτά τα οποία ε, ήδη ελέγχθησαν. Γιατί το πότε τώρα δεν χρειάζεται αυτό. Πάντως ευχαριστούμε την κύριε Επίτροπο για την πρωτοβουλία και για την άμεση αντίδραση και θεωρώ ότι ε, και εμείς μπορούμε να δεσμευτούμε ότι θα είμαστε ε, διαθέσιμοι και ότι θετικά θα διακύμεθα προς την πρότασή σας. Και από πλευράς ε, ε διεκπαιρέωσης αλλά και από πλευράς συμφωνίας με τις λεπτομέρειες και τα ποσά τα οποία ε, περιέχονται στην πρότασή σας. Οπότε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα και θα πρέπει να προσθέσουμε κάτι, θα πρέπει να διευκρινίσουμε, θα πρέπει να ε, διαφωνήσουμε, όπως τα είπε ο κ. Ντεπρέ. Και πάντως, πέραν αυτών, ήθελα να σας πω ότι η Frontex θα πρέπει να έχει ξεκάθαρη ρότα σε αυτή τη στιγμή. Οπότε και το Κοινοβούλιο είναι διατεθειμένο να την ενισχύσει ακριβώς. Θα πρέπει να δούμε και τι προβλέπεται να γίνει και τι προοικοδότηση προβλέπεται να υπάρξει. Οπότε θα πρέπει να συμφωνήσουμε, δεν είμαι τόσο σίγουρος να συμφωνούμε σε σχέση με αυτά που έχει προτείνει το Συμβούλιο. Είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Χρειάζονται πράγματα τα οποία προηγουμένως δεν είχαν ανακύψει. Άρα και εμείς θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε, να καλύψουμε αυτές τις νέες ανάγκες χωρίς να επιστρατεύσουμε φρέσκους πόρους, φρέσκα χρήματα. Να τετραγωνίσουμε τον κύκλο, να τα καταφέρουμε όλα χωρίς να προσθέσουμε μια δεκάρα αυτό πολλές φορές τελικά καταλήγει να θέτει εν κινδύνο το σύνολο της ισορροπίας του προϋπολογισμού. Έχουμε το μέσο ευελιξίας, ε, θα πρέπει να δούμε πόσο και πώς θα χρησιμοποιηθεί, οπότε όλα αυτά θα ξεκαθαριστούν καθώς θα αποκρισταλώνεται η τοποθέτησή μας. Τώρα τελευταίο κύριε Επιτροπέ, έχω την εντύπωση ότι δεν μπορούμε παρά να ακολουθούμε τα γεγονότα και να αντιδρούμε εκ των υστέρων και πάλι καλά. Όμως νομίζω ότι ε, τη σήμερα ημέρα έχουμε όλα τα στοιχεία, όλες τι πληροφορίες για να μπορέσουμε να προλάβουμε τις ε, εξελίξεις όλα αυτά τα οποία επιβάλλονται. Και μιλώ όχι μόνο για τους υπόλοιπους μήνες του 2015 αλλά και για το 2016 να έχουμε ένα πρώτο σχέδιο για το 2016. Αλλά δεν είμαι σίγουρος για το ότι ε, είμαστε έτοιμοι, έχουμε καλύψει αυτά τα οποία και εσείς μας λέτε για το 2016. Όλα αυτά που θα απαιτηθούν για το 2016. Πάντως, σε αμέσως επόμενες εβδομάδες και με τη συνδιαλλαγή θα μπορέσουμε να δομήσουμε αυτή μας την ε, ε, ικανότητα πρόληψης. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Λόγω στον κύριο Τζάνι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την κυρία Επίτροπο που για άλλη μια φορά έδειξε το πόσο είναι διατεθειμένη να βοηθήσει την Επιτροπή μας. Οπότε θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοι να δούμε το πώς θα υλοποιήσουμε αυτά τα κατεπήγοντα μέτρα. Να την ευχαριστήσουμε και πάλι. Και ξεκινώ με αυτό που στο τέλος ανέφερε ο κύριος Μαραγκάλ. Πάρα πολύ ε, εύστοχο είναι η διορθωτική σας πρόταση, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα για μια δέσμη μέτρων που δεν έχει να κάνει μόνο με την δική μας Επιτροπή για αυτή την κατάσταση των ανάγκης, αλλά χρειάζεται μια δέσμη μέτρων ευρύτερη που να κάνει κάτι για τις αιτίε του προβλήματος. Είδαμε τι γίνεται με όλους αυτούς που φτάνουν στην ε, Γερμανία. Μιλάμε για 9-10 άτομα την ημέρα και έχουμε το 15 ε, εκατοντάδες χιλιάδων που θα έχουν φτάσει. Και επομένω όλα αυτά τα νούμερα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά και δεν νομίζω ότι τα κατεπήγοντα μέτρα του προηγούμενου του 15 πρόκειται να καλύφθουν τις ανάγκες του 16 που έχουμε τον άλλο προπολογισμό. Γιατί θα πρέπει να δούμε πώς θα είμαστε πιο συντονισμένοι, Κομισιόν και Κοινοβούλιο και πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο που όπως έχουμε δει είναι δύσκολες όσον αφορά ε, αυτές τις 120.000 που προβλέπεται να κατανεμηθούν και πόσο αυτό το σχετικά μικρό νούμερο έχει δημιουργήσει στα κράτη-μέλη. Τώρα θέλω να σας τονίσω και κάτι άλλο, το οποίο δεν τονίστηκε από τους προελέξαντες συναδέλφους όσον αφορά τον έλεγχο για αυτούς τους πόρους. Είναι σημαντικό να εκταμευτούν αυτά, είναι σημαντικό να συμβάλλει ο κοινωνικός προϋπολογισμός. αλλά το θέμα είναι το ότι δεν θα πρέπει να επιβαρυνθούν τα κράτη-μέλη που για γεωγραφικούς λόγους είναι κοντά στην είσοδο αυτών των μεταναστών, αυτών των ροών, γιατί θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί με τον έλεγχο. Ξέρουμε πόσο δυσκολεύεται η Όλαφ όσον αφορά τον έλεγχο της ε, ορθής αξιοποίησης των ε, πόρων. Ε, όταν επισημαίνεται κάποια ενδειχόμενη απάτη, απευθύνει στο κράτο μέλο η Όλαφ και το κράτο μέλο λέει το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η Όλαφ αργότερα. Να, έγινε αυτό και με την Ιταλία, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται στι άλλε χώρε τη Ένωση. Και σε επαφέ με τα Υπουργεία είδαμε ποιε είναι οι δυσκολίε όσον την αξιοποίηση αυτών των ε, πόρων. Οπότε θα πρέπει να καταβληθεί μια επιπλέον προσπάθεια και από την κυρία Επίτροπο και από την ε, Επιτροπή μας, τόσο ώστε να υπάρχει περισσότερος έλεγχος για αυτούς τους ε, πόρους και πώς αξιοποιούνται. Αλλιώς θα, δεν θα πρέπει να ε, έχουμε βιαστική συμπεριφορά και να ακολουθούμε τις εξελίξεις γιατί ακριβώς δυσκολευόμαστε να επέμβουμε επί τόπου και επομένως χρειάζεται μια παραπάνω προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος, σύμφωνα με τον κύριο Τζάνι, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος και θα πρέπει να προλαβαίνουμε κάθε εκτροπή. Αλλά είδαμε στην Ιταλία, όπου πήγα και στην Σικελία συγκεκριμένα. Οπότε η πρώτη μου εντύπωση ήταν ότι η ευρωπαϊκή πόροι ήταν απλώς το 10% των ε, δαπανών της κυβέρνησης και των τοπικών αρχών της Ιταλίας. Οπότε, πόσο να πιέσουμε ως Ευρώπη, ως Κοινοβούλιο. Θα δώσω πρώτο λόγο στην Γενική Συγκεντρία και στους συντονιστάς και βεβαίως και στους συναδέλφους. Και όμως αυτούς τους ε, πόρους που απορρέουν από τον προϋπολογισμό ή από τα παραρτήματα, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, κάτι το οποίο γίνεται τον προϋπολογισμό, το οποίο τροφούνται από τα κρατή-μέλη, οπότε άμεσα εκεί συμφέρουν τα κρατή-μέλη και θα, θα πρέπει αν μπορέσετε να μας δώσετε μια εικόνα του τοπίου γενικότερη τι γίνεται το 2015 ή το 2016, τι γίνεται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη, τι γίνεται με αυτέ τι ε, εισφορέ των κρατών μελών, για να δούμε γιατί, τι γίνεται με την αποτελεσματικότητα των ε, σκοπουμένων μέτρων και να δούμε πώ θα έχουμε απλούσταση των διαδικασιών και περισσότερη αποτελεσματικότητα. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Είναι πολύ ε, σημαντικά και ενδιαφέροντα τα ερωτήματα και θα προσπαθήσω να δώσω τις καλύτερες δυνατές απαντήσεις, αναγνωρίζοντας ε, βέβαια ότι με τις λεπτομέρειες θα καταλάβετε κι εσείς καλύτερα και θα μπορέσουμε και εμείς να απαντήσουμε και σε άλλα ερωτήματα που τυχόν προκύψουν. Συμφωνώ απόλυτα με τον πρόεδρο Βαρτουή ότι έχουμε δει πόσο σημαντική είναι η ευελιξία κρίσης. Έτσι εστιάζουμε λοιπόν ακόμα πιο πολύ στον προϋπολογισμό που πρέπει να είναι ένας προπολογισμό ε, που θα προσφέρει πλήρως τις υπηρεσίες του στην Ευρώπη και θα εμβαθύνει την ευελιξία. Ας ε, προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα όπως μετέθησαν. Καταρχάς, σχέση μεταξύ ανλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να καλύψουμε εν μέρει τις πληρωμές λόγω της πιο αργής από ό,τι περιμέναμε υλοποίηση ε, προγραμμάτων συνοχής και άλλων προγραμμάτων. Πρέπει όμως ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε ότι μέρος των πληρωμών θα πρέπει να καταβληθεί εντός του 16 και πολύ σωστά είπατε αυτό σημαίνει ότι όταν καταθέσουμε την πρότασή μας για την τροποποίηση του προπολογισμού του 2016 θα πρέπει να δίνουμε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Ε, Επίση, ε, ρωτήσατε συγκεκριμένα για τα 170 εκατομμύρια. Είναι, ε, θα έλεγα και μεγαλύτερο τελικά αυτό το ποσό. Έχει να κάνει με το Global Transfer, τη συγκεντρωτική μεταφορά υπολείπου. Εκεί εντάσσεται. Σε 47 κονδύλια του προπολογισμού θα γίνει με ίτερ 97 εκατομμύρια και Κοπέρνικους 53 εκατομμύρια ε, τα κονδύλια που συνεισφέρουν περισσότερο. Αλλά έχουμε και άλλε 45 γραμμές του προπολογισμού. Ουσιαστικά κοιτάξαμε πρόγραμμα, ε, ε, με πρόγραμμα, κονδύλιο με κονδύλιο για να δούμε από πού μπορούμε να αντιλήσουμε την μέγιστη χρηματοδότηση. Και για να ελαφρύνω λίγο ε, το κλίμα, να σας πω ότι οι συνάδελφοί μου στην ε, Κομισιόν θα με λένε κρυσταλλίνα η σκούπα. Διότι πραγματικά ε, σκούπισα και ξεσκόνησα ε, τα πάντα για να βρω και το τελευταίο σέντ διαθέσιμο. Κάτι άλλο το οποίο με ρωτήσατε ήταν πώς αυτό το, αυτά τα ποσά, η χρηματοδότηση ε, πώς υποδιορείται στο 15 και στο 16. Λοιπόν, το 2015 προτείνουμε 950 εκατομμύρια από τα 2,9 δις του επιπλέον αυτό ποσό που σας ε, περιέγραψα. Το 2016 1,95 δις ευρώ. Τόσο σε αφορά συνολικά να σας πω, ξεκινήσαμε το έτος με 4,5 δις. Ήταν στον προπολογισμό του 15 και του 16 το ποσό αυτό. Προσθέσαμε με δύο προτάσεις της Κομισιόν 1,2 δις και 1,7 δις για τις κατηγορίες 3 και 4. Και αυτά τα 2,9 δις που μεταξύ του 15 και του 16 όπως σας είπα, 950 εκατομμύρια πηγαίνουν το 15 και 1,95 το ε, δις το 16 και έχουμε πάρει χρήματα κυρίως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, ναι. 1,8 δις Trust Fund για την Αφρική. Άρα, συνολικά φτάνουμε σε 4,7 δις παραπάνω Άρα πάνω από τα διπλά σε σχέση με τα χρήματα με τα οποία ξεκινήσαμε. Αυτό συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ τελικά να απαντήσω στις ερωτήσεις με τη σειρά. Θα κάνω μια σύνθεση ε, στις απαντήσεις μου. Ένα πολύ σημαντικό σημείο ήταν ότι θα πρέπει να είμαστε πιο διορατικοί και όχι απλά να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Εγώ θέλω να τονίσω και για τη δική μου ομάδα και για την Επιτροπή ότι όταν παρουσιάσαμε το σχέδιο προεμβολισμού του 2016, πριν χτυπήσει αυτή η κρίση, είχαμε προτείνει πολύ σημαντικές αυξήσεις σε τρεις τομείς. Μετανάστευση, 30% αύξηση σε σχέση με το 2015 στην κατηγορία 4, εξωτερικές δράσεις, 28,5% αύξηση σε σχέση με το 2015 και βέβαια Ανάπτυξη απασχόληση περίπου 30% αύξηση. Με άλλα λόγια. Το είδαμε να έρχεται. Βέβαια δεν ε, είχαμε προβλέψει ε, τις διαστάσεις, το μέγεθος του προβλήματος, αλλά το βλέπαμε να έρχεται. Και πραγματικά ε, το είδαμε και στην πράξη. Το θέμα είναι βέβαια να ακολουθούμε σωστές προτεραιότητες. Υπάρχει ένα ερώτημα για το βαθμό στον οποίο πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τις απαιτούμενες πληρωμές και να κάνουμε πράξη αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε πράξη. το μηχανισμό ευελιξία, αλλά χωρί να ξεπερνάμε τα ανώτατα όρια στην οροφή. Εμεί στην Κομισιόν πιστεύουμε ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, κατανοεί ότι ο μηχανισμός ευελιξία πρέπει να είναι εκτός πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και εκτό εκτός οροφών. Δεν υπάρχει όμως ακόμη ε, κοινό έδαφος με το Συμβούλιο. Θα το συζητήσουμε όμως αυτό. Στην διάμεση αναθεώρηση θα έχουμε χρόνο να τα δούμε όλα αυτά τα ζητήματα. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω μια σημαντική έκκληση ότι πρέπει να δούμε με τη σειρά τα πράγματα. Πρώτα πρέπει να κινητοποιήσουμε αυτούς τους πόρους, να τους αξιοποιήσουμε. Ελπίζω λοιπόν να μην είναι όμοιρος αυτή η επίγουσα δράση μας ε, στην προσπάθεια επίλυσης πιο μακροπρόθεσμων προβλημάτων. Που ναι υπάρχουν, ναι πρέπει να επιληθούν, αλλά σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη πρόταση ελπίζω να μην κολλήσουμε στο αν είναι πάνω ή κάτω από την οροφή. Έχουμε τα χρήματα μπορούμε και για φέτος και για το 2016 να τα διαθέσουμε Παναλαμβάνω κυρίως λόγω του ότι ε, δεν απορροφήθηκαν στον βαθμό που θα, θα, είχαμε, που θα περιμέναμε τα κονδύλια. Το Ταμείο Συνοχής για τον περιπολισμό του 2016 τώρα θέλουμε στοιχεία για τη γεωργία, πιο αναλυτικά στοιχεία και μετά θα δώσουμε τα οριστικά νούμερα. Χρειάζεται λοιπόν λίγος χρόνος ακόμη. Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου θα είμαστε έτοιμοι. Τι θα κάνουμε ακριβώς με αυτά τα χρήματα ήταν ένα ερώτημα για τις τρίτες χώρες συγκεκριμένα από τι οποίε φεύγει ο κόσμο. Έχω την τιμή να έχω αναλάβει ε, αυτό το έργο κατά το παρελθόν ε, και έχω πάρα πολλά στοιχεία να σας δώσω. Πρέπει να σας πω ότι συνδυάζομαι την ανθρωπιστική βοήθεια και πόρους από τα μέσα γειτονία. Για τρία πράγματα κυρίως. Πρώτον, να αντιμετωπίσουμε τις άμεσες ανάγκες επιβίωσης, δηλαδή φαΐ, στέγη. Δεύτερον, να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες, τις πιο μακροπρόθεσμες, που είναι και αυτές όμως πάρα πολύ σημαντικές, δηλαδή εκπαίδευση και ε, υγειονομική περίθαλψη. Για τα παιδιά των προσφύγων και των μεταναστών, υγειονομική περίθαλψη. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από μια οικογένεια το να βγάλει τα παιδιά της από το σχολείο και να μην υπάρχει πια καμιά προοπτική για αυτά τα παιδιά να γίνουν παραγωγικά ε, στελέχη της κοινωνίας. Για την Ιορδανία, για το Λίβανο και για την Τουρκία ακόμη, τα σχολεία ε, είναι τόσο γεμάτα που τα παιδιά δεν μπορούν να, να φοιτήσουν. Το συζητήσαμε και με τον Κόρτον Μπράουν για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των παιδιών των προσφέρων Ξεκινήσαμε και με το τον λέει και με τη UNICEF No Lost Generation να μην υπάρχουν χαμένες γενιές έτσι λεγόταν το πρόγραμμα πριν από κάποια χρόνια και σίγουρα πρέπει να ε, παραμείνουμε εστιασμένοι σε αυτό γιατί αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη απόγνωση στους γονείς και ε, τους διώχνει από τις χώρες τους όταν δεν μπορούν δηλαδή τα παιδιά τους να πάνε σχολείο. Φυσικά και θα πρέπει να δούμε και δύο χρόνια, τρία μπροστά μας ε, τι περιμένουμε να γίνει. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης για όσους φεύγουν και από το πόλεμο στη Συρία κυρίως, αλλά και από άλλες ε, προβληματικές περιοχές. Με ρωτήσατε επίσης κατά πόσον αναμένουμε ότι θα πρέπει να γίνουν νομοθετικές αλλαγές ή προσαρμογές. Ναι, σε δύο επίπεδα. Πρώτον, για τις επιστροφές και είπατε θα χρηματοδοτηθούν οι επιστροφές με μέρος των κονδυλίων. Θα πρέπει να το δούμε πιο συγκεκριμένα. να έχουμε μια ε, διαφορετική μεταχείριση για αυτούς που πραγματικά φεύγουν από τους διωγμούς και από τους πολέμους σε σχέση με αυτούς που έρχονται στην Ευρώπη αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Φυσικά η φιλοδοξία είναι θεμητή, μιλάω για τη δεύτερη κατηγορία ανθρώπων, αλλά δεν θα δώσουμε σε αυτούς προτεραιότητα τουλάχιστον στην παρούσα χρονική στιγμή. Φυσικά, αυτοί οι οποίοι έρχονται αναστώντα μια καλύτερη ζωή, αν υπάρχουν δουλειέ για αυτούς, όλα καλά. Αν δεν υπάρχουν όμως, ως Ένωση θα πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα, να είμαστε πιο πειθαρχημένοι και να βοηθήσουμε πρώτα απ' όλα αυτού που θα επιστρέφουν. Και όταν επιστρέφουν, Θα πρέπει και την αναπτυξιακή πολιτική και τη σχετική χρηματοδότηση να την συνδυάζουμε με αυτή ε, τη δράση επιστροφής αυτών των ανθρώπων στις χώρες για να μπορούν να βρίσκουν εκεί δουλειά. Πίσω στις πατρίδες τους. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι δεν το είδαμε τόσο σοβαρά το ζήτημα αυτό της ευθυγράμμισης δηλαδή της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής πολιτικής με τις νέες πραγματικότητες του κόσμου που είναι πιο εύθραυστος, που έχει περισσότερε κρίσει. Έχουμε το θεματολόγιο για την ε, αλλαγή και την ανάπτυξη. Εστιάζουμε δηλαδή σε πιο έφραστες χώρες, σε πιο ευάλωτες χώρες, αλλά πρέπει να εστιάσουμε ακόμη περισσότερο στην πιο καλή ανάπτυξη ε, της πολιτικής της Ένωσης και της διάθεσης των κονδύλων για να έχουμε ισορροπημένες δράσεις. Δεν αρκεί να γυρίζουν πίσω κάποιοι άνθρωποι αν δεν έχουμε εξασφαλίσει το τι θα συμβεί ε, σε αυτούς τους ανθρώπους όταν γυρίσουν πίσω στις χώρες τους. Η δεύτερη νομοθετική δράση που έχουμε μπροστά μας είναι να ορίσουμε πώς θα προστατεύσουμε τα σύνορα της Ένωσης. Και σίγουρα πρέπει να γίνουν πράγματα σε αυτό το μέτωπο. Με ρωτήσατε αν για τον ΕΑΣΟ για τη Europol και το Frontex προτείνουμε ε, αύξηση αυτών των μέσων μόνο για φέτος. Φυσικά και όχι, δεν νομίζω ότι θα έχει ολοκληρωθεί, δεν θα έχει περάσει η κρίση. Είμαστε εκτός του, της 5% εδώ. Φυσικά με τέτοιες προτεραιότητες όπως αυτή θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια μεσοπρόθεσμη προοπτική Εντάξει, έχουμε δεσμευτεί για αυτό το 5% μείωση. Θα το δούμε πιο μεθοπρόθεσμα γιατί πρέπει τώρα να δούμε τι είναι πήγον και τι είναι κρίσιμο. Εξετάζω ακόμη τις ερωτήσεις που με έχετε θέσει. Σχετικά με την ποιότητα των ελέγχων. Κυρίως όταν κάνουμε κινήσεις, μετακινούμε με ανθρώπους με μεγάλη ταχύτητα. Το έχουμε αυτό τώρα στο ραντάρ μας και ε, έχει μεγάλη σημασία να ξανασκεφτούμε ολόκληρη ολόκληρο τον στόχο των διαφόρων μέσων. Για παράδειγμα, ανθρωπιστική βοήθεια. Εξορισμού. Η δράση αυτή πρέπει να είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανθρωπιστική βοήθεια δίνουμε καταρχήν σε φτωχές χώρες. Όμως, βρισκόμαστε πραγματικά σε εντελώς έκτακτες καταστάσεις. Ήδη κάναμε μια εξαίρεση και δώσαμε ανθρωπιστική βοήθεια στην Ιαπωνία μετά από την καταστροφή που υπέστη πριν από λίγα χρόνια. Και το ερώτημα τώρα είναι, ακολουθούμε τις χώρες ή ακολουθούμε τους ανθρώπους. Αν έχουμε εκατομμύρια μεταναστών ή μάλλον προσφύγων που έρχονται στην Ευρώπη. Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν πρέπει να εφαρμοστεί, δεν πρέπει να δοθεί τέλος πάντων σε αυτούς, δηλαδή πρέπει να ακολουθήσει τις ανάγκες των ανθρώπων αυτών. Προφανώς δεν πρόκειται να λύσουμε το θέμα αυτό σήμερα, αλλά απλώς σας, δείχνω, δίνω ένα παράδειγμα μια ευρύτερη άποψη. Δηλαδή πρέπει να επαρεξετάσουμε του μηχανισμού που διαθέτουμε. Αναφύονται νέε πραγματικότητε και πώ μπορούν να ευθυγραμμιστούν οι μηχανισμοί μα με τι πραγματικότητε που αναφύονται. Ελπίζω να απάντησα σε όλε και όλου. Μήπω ξέχασα κάτι. Αν ναι, οι συνάδελφοί μου εδώ μου λένε, αν μου υπενθυμίζουν κάτι, ίσως να είναι αυτονόητο, αλλά ας το πω. Είναι κατεπίγουσα η κατάσταση. Επομένω, ας προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ο πρόεδρος Αρτουή θα αναμείνουμε και την ε, απάντηση του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κυρία ε, Επίτροπη για τις απαντήσεις σας. Θα δώσω το λόγο ε, στις και στους συναδέλφους μας εκείνους που επιθυμούν ακόμη να τοποθετηθούν. Ο κύριος Μπέγκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την κυρία Επίτροπο που ευθύς αμέσως την λήψη αποφάσεως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσήλθε ενώπιόν μας. Και μου φαίνεται καλό που στο τέλος της παρεμβάσεώς της υπενθύμησε και πάλι την αναγκαιότητα να δοθεί βοήθεια κατεπηγόντως και χωρίς να λησμονούμε ότι χρειαζόμαστε και βραχυπρόθεσμα μέτρα σταθεροποίησεως και στρατηγικό προβληματισμό της διεθνούς κοινότητας για το πώς ποια θα είναι τα επόμενα βήματα εφόσον πρόκειται να κάνουμε και κάποια ανοικοδόμηση των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι πρόσφυγες. Δεν λέμε ότι τα πράγματα αυτά είναι κατεπήγοντα. Δεν μπορώ ωστόσο να αποφύγω να πω ότι προφανώς δεν διαθέτουμε ούτε σε διεθνές επίπεδο, ούτε σε παγκόσμιο επίπεδο, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν διαθέτουμε τα μέσα και τους μηχανισμούς για να μπορούμε να ανταποκρινόμεθα άμεσα. Ας εξετάσουμε τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά και τον προπολογισμό της Ομοσπονδιακής Γερμανίας, της πατρίδας μου αλλά και τον προπολογισμό των περισσότερων άλλων χωρών μελών που παρόλη την, παρόλο το κατεπήγον της καταστάσεως μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου είχαν διαθέσει μόλις το 40-50% των κονδυλίων που είχαν υποσχεθεί για το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Διατροφής. Ήδη εσείς, στα τέλη Σεπτεμβρίου, στην ανακοίνωσή σας, τονίζετε και δικαίως ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων για την Συριακή κρίση από τα 4 περίπου δισεκατομμύρια που εκτιμάται ότι χρειάζονται έχουν φτάσει οι διαθέσεις κονδυλίων μονάχα το 38% και μετά στην ίδια ανακοίνωση προτείνεται 2 δισεκατομμύρια από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, από τον, Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και από τις χώρες μέλη να οδεύσουν προς τα εκεί. Να μην λησμονήσουμε ότι το να μην αναλάβει δράση κανείς στο κατάλληλο χρονικό σημείο, αυτή η παράληψη δράσης έδωσε ακόμη μια γυρίσπροξιά προξιά σε, αυτή, σε αυτό το προσφυγικό κύμα. Γι' αυτό λοιπόν και είναι απολύτως κατεπήγον να αντιδράσουμε ταχύτατα και να φτιάξουμε μια σωστή δέσμη. Και απευθύνομαι και στο Συμβούλιο Υπουργών. Και παρακαλώ να μεταφερθεί το μήνυμα. Στην πρώτη ανάγνωση 2.16 η στάση του Συμβουλίου θα έλεγα ήταν γελία αν δεν ήταν τόσο δραματική κατάσταση. Όμως το Συμβούλιο θα κληθεί να απαντήσει και σε σημαντικά ερωτήματα. Εάν τώρα κυρία Επίτροπε αυτό το Transfund για την Αφρική το οποίο προτείνεται και στο οποίο κάνετε σημαντικές μεταφορές. Εκεί υπάρχει και μια γραμμή που λέει συνεισφορές των χωρών μελών. Μόνο η Ισπανία και η Γαλλία έχουν δηλώσει διατεθειμένες να δεσμευτούν. Μιλήσατε και για το Ταμείο της Ελπίδας. 1,8 δισεκατομμύρια. Δύο χώρες έχουν κάνει κάποια συνεισφορά στο Ταμείο αυτό, σε πολύ χαμηλό επίπεδο, η Ιταλία και η Γερμανία μόνο. Και κάποια χρήματα από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Το έρχεστε και ξαναπροτείνετε 300 εκατομμύρια από το ΕΝΠΗ και 200 εκατομμύρια από το πρόγραμμα προενταξιακών ενισχύσεων και άλλα 500 εκατομμύρια ελπίζεται ότι θα προέλθουν από τις χώρες μέλη, έτσι ώστε να δείξουμε ότι ανταποκρινόμαστε στις υποχρώσεις μας. Αυτό λέτε. Κατανοώ βέβαια ότι είστε υποχρεωμένοι να προσφύγετε σε αυτά τα μέσα, διότι δεν υπάρχει πραγματική ευκαιρία να καθίσουμε να συζητήσουμε ειλικρινώς για τα όσα μας απασχολούν και τώρα και για το επόμενο χρονικό διάστημα ότι χωρίς μαζική αναθεώρηση τη δημοσιονομική προοπτική δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Τώρα θέλω εγώ να δω πότε θα είναι σε θέση οι χώρες μέλη και το Συμβούλιο Υπουργών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσει του, να καλύψουν τις, παραλύσεις τους, τις παραλήψεις τους. Βεβαίως πάντα με τα τέλη του έτου, οι συνεισφορέ μεγαλώνονται λίγο παραπάνω. Αλλά μέχρι τώρα φοβόντουσαν. Όποιο πιάσει τον Μικάδο στο παιχνίδι αυτό με τα ξυλαράκια, όποιο δεν θα, θα χάσει. Όποιο κάνει την πρώτη κίνηση δηλαδή. Λέτε τώρα τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο για κατεπήγοντα. Και στο επίπεδο των G7 και άλλων χωρών λέτε, λένε μάλλον ότι θα διαθέσουν 1,8 δισεκατομμύρια Επίσης 560 εκατομμύρια για τα οποία είχε δεσμευτεί η κυρία Μογκερίνη αρχές του έτους. Είναι σημαντικά τότε αυτά που είπε ο κ. Σαρτουή, ότι σιγά σιγά αρχίζει και προκύπτει μια σύγχυση στα νούμερα. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο να μας διατεθεί ένας ξεκάθαρος κατάλογος όλων των κονδυλίων για να μπορούμε να συζητούμε και καθαρά. Το, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να απευθύνω έκκληση στο Συμβούλιο να προχωρήσει ταχύτατα και όχι μονάχα να λαμβάνει δεσμεύσεις και να δίνει διαβεβαιώσεις αλλά και να πει καθαρά πότε θα εκρέψουν τα κονδύλια. Και ήδη είναι καθυστερημένο. αυτό που γίνεται εδώ είναι ο πραγματικό έσχος. Και θα φορτωθείτε το κρίμα ότι θα έρθει άλλο ένα εκατομμύριο πρόσφυγες στην Ευρώπη διότι δεν αντιδράσατε έγκαιρα. Με τις παρατηρήσεις μου αυτές, κυρία Επίτροπε, δεν αμφισβητώ βεβαίως την ταχύτητα των αποφάσεων σας και βεβαίως πρέπει να καταπιούμε και κάποια πράγματα όπου δικαίως θέτουμε το ερώτημα. Τα μακροπρόθεσμα μέτρα σταθεροποιήσεως που είναι απαραίτητο να ληφθούν, πώς θα ληφθούν όταν τώρα πηγαίνω και παίρνω από τα τρία προγράμματα γειτονίας όπου ούτω ή άλλω το Συμβούλιο έχει προβλέψει 450 εκατομμύρια περικοπέ, να έρθετε να μα πείτε ότι παίρνω λίγα λεφτά από εδώ, λίγα λεφτά από εκεί. Αντιμετωπίζουμε και την Τουρκία, η οποία αναγκάστηκε να δεχτεί περικοπέ των κονδυλίων που λαμβάνει κατά 176 εκατομμύρια και μιλούμε για τέτοιε μεταφορέ για να χρηματοδοτήσουμε τα μέτρα αυτά. Έχετε δίκιο ότι το ζήτημα ουσία πρέπει να τεθεί. Τι κάνουμε με τα διεθνή μας προγράμματα, όπου περιλαμβάνεται και η δημοσιονική βοήθεια, βοήθεια που δίνεται για συγκεκριμένα προγράμματα και ούτω καθεξής. Και βεβαίω και για την Αφρική και τη συνεργασία μας με τις χώρες της Αφρικής για ανάπτυξη. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι περικόπτουμε κάποια χρήματα από κάποια αναπτυξιακά προγράμματα για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε το Ταμείο της Ελπίδας και όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε με την ησυχία μας. Εάν συμφωνήσουμε με τις μεταφορές αυτές πιστώσεων, τότε αναμένω σε μια επόμενη φάση, και εσείς κύριε Επίτροπε και οι υπόλοιποι Επίτροποι, να καθίσετε να προβληματιστείτε ποια πράγματα είναι απαραίτητα για να προκύψει μια σταθεροποίηση και πώς θα πρικοδοτηθούν τα προγράμματα αυτά για να μην ξαναπέσουμε σε μια τρύπα και απολεστεί οριστικά και τελεσίδικα πλέον η αξιοπιστία μας. Γι' αυτό η παράκλησή μου είναι να εγκύψετε στο θέμα αυτό όσο το δυνατόν ταχύτερα, διότι ήδη έχουμε φορτωθεί πολλές ευθύνε. Γιατί μέχρι τώρα κινούμαστε με την ταχύτητα σαλιγκαριού. Και μια τελευταία παρατήρηση. Όταν θα εξομαλυθούν λίγο τα πράγματα, πρέπει να συζητήσουμε λίγο τους μηχανισμούς που διαθέτουμε. Γιατί άλλο πράγμα είναι η νομοθετική εργασία και άλλο είναι η ταχύτητα των αντιδράσεων. Πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε να εφαρμόσουμε διαδικασίες fast track. Εκεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες μέλη πρέπει να κουράσουν λίγο την ε, θεά τους ουσία. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ κύριε Μπέργκε. Ο κύριος Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Πρώτα πρώτα, ευχαριστούμε που ήρθατε και ελπίζουμε αυτό να επαναληφθεί. όχι βέβαια ε, για κάποιους καταστάσεις, αλλά τόσο για να έχουμε κάποια ενημέρωση, ανακοίνωση, γιατί μας παίρνετε στα σοβαρά και το οποίο δεν είναι αυτονόητο. Οπότε ευχαριστούμε. Τώρα, μία ερώτηση πολιτική υφή γιατί παρατηρήσει τον προπολογισμό. Η παρατήρηση είναι ότι έχουμε του συναδέλφου μα στην ΑΦΕΤ που μα ενημέρωσαν ότι ένα από του λόγου ε, αυτή τη μαζική ροή μεταναστών είναι το ότι έχουν συρρυκνωθεί τα κεφάλαια τα οποία χορηγούνται σε Τουρκία και Λίβανο στρατόπεδα μεταναστών και προσφύγων. Επομένω, για πετε μα, ποιο έκανε αυτέ τι περικοπές και τι ύψου είναι. Δεν ήταν τα χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και λένε σήμερα οι πολιτικοί αυτοί ότι αυτό είναι από του λόγου τη μαζική εισρωή. επομένω, ποιο είναι ο ένοχος. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αλλά προσπαθώ να καταλάβω πώς έχει η κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δοθούν πίσω τα χρήματα και έτσι να αρθεί αυτό το κενό χρηματοδότησης ή υπάρχει κάτι καινούργιο. Αυτό από πολιτικής πλευράς, τώρα από δημιουργικής. Η κυρία Γκάρτια η κυρια γκαρδια θαμπαλ σας ερώτησε κάτι για πιστός πληρωμών και υποχρεώσεων και αυτά τα περίφημα ανεξόφλητα, το backlog δεν ξέρω αν συνεχίζει να ισχύει το πρόβλημα αυτό, αλλά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα γιατί έχουμε πρόταση για τον χρόνο 2%. Ακόμα και με την επιβράδυνση της συνοχής με τις νέες ταπάνες, αυτό είναι σκαμπανάκι κινδύνου. Οπότε ας το πούμε ανοιχτά, ότι θα είναι δύσκολο να κάνουμε κάτι για τα ανεξόφλητα και θα έχουμε περισσότερα τις επόμενες χρονιές. Και ε, άλλες δύο ερωτήσεις. Θέλω κύριε Επιτροπέ τη γνώμη σας. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της συνδιαλλαγής και συγκεκριμένα όσον αφορά την αναθεώρηση του πολίτου δημοσίου πλαισίου και όταν προτείνεται αυτή την αναθεώρηση Αυτό θα πάει για το τέλος του έτους ή για Απρίλιο-Μάιο. Συγγνώμη που αυτό το λέω προεξαγγελτικά πριν ληφθεί απόφαση, αλλά είναι όλο ένα και πιο σημαντικό για μας. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Κυρία Χολμάιρα. Πρώτα, συμφωνώ απολύτως με τον τα συνάδελφό μου Μπέγκε. Τα ίδια με απασχολούν και εμένα. Οι αποφάσεις που λάβαμε τους τελευταίους μήνες νομίζω ότι δεν εξυπηρετούν την διαχείριση και αντιμετώπιση ούτε και πρόβλεψη των κρίσεων ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στις χώρες μέλη. Θεωρώ ότι τα πήγαμε πολύ άσχημα. Αγνοούμε τις αναφιόμενες εξελίξεις μέχρι ότου αυτές να μας χτυπήσουν κατά πρόσωπο. Και τότε αναγκαζόμαστε να τις αντιμετωπίσουμε με λύσεις ανάγκης. Τα όσα μας εξηγήσατε τα, τα, ε, τα βλέπω θετικά και θα προσπαθήσω να σας υποστηρίξω. Όμως, με ενδιαφέρει και η μεσοπρόθεσμη προοπτική. Μεσοπρόθεσμα. Μέχρι πότε θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξηγήσει τι θα κάνει τα επόμενα 2, 3, 4 χρόνια. Πώς θα αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή για τα επόμενα χρόνια. Αν δεν έχουμε κανένας είδους πρόγνωση. Το πρόβλημα που έχουμε με την κρίση του, των προσφύγων δεν πρόκειται να τελειώσει σύντομα. Θα αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα και για τα επόμενα δύο και τρία χρόνια. Η ερώτησή μου είναι έχετε υπόψη κάποιο χρονοδιάγραμμα. Έχει αντιληφθεί την ανάγκη αυτή το Συμβούλιο. Εξετάζοντας τα κονδύλια της πολιτικής γειτονίας, από την Τουρκία προέρχονται οι περισσότεροι πρόσφυγες. Θα πρέπει να στηρίξουμε την Τουρκία περισσότερο και σε μεγαλύτερη διάρκεια. Τώρα με ποιον τρόπο βέβαια πρέπει να συζητηθεί ακόμη. Για τα όσα μας είπατε, έχω μία συγκεκριμένη ερώτηση. Ο πρόεδρος διακόπτη. Παρακαλώ, όσο γίνεται συντομότερα, γιατί στις 12.30 ακριβώς είναι υποχρεωμένη να αποχωρήσει η κυρία Επίτροπος. Πρώτα σε, πρώτη, εμένα απευθύνεται την έκκληση αυτή κύριε Πρόεδρε. Αλλά καλώς. Να συνεχίσω όμως και τέλειως Ερώτηση λοιπόν για το αποθεματικό για την βιώσιμη αλία. Μείον 18 εκατομμύρια. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να υποστηρίξει χώρες της Βόρειας Αφρικής για παράδειγμα για να διαχειρίζονται με πιο βιώσιμο τρόπο την αλία τους. Μην πάμε τώρα να ρίξουμε κάποιους άλλους στην δυστυχία, προσπαθώντας να απαλύνουμε την δυστυχία άλλων. Και τα μείον 2,2 εκατομμύρια στην ε, citizenship και ασφάλεια της ηθαγένειας, αυτό δεν το κατανοώ. Τέλος, νομίζετε ότι οι πληρωμές που σχεδιάζουμε για το 2016 θα αρκέσουν για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες μέλη. Ασφαλώς όχι, κύριε Πρόεδρε Εσείς, κύριε Αλίεφ. Ε, λοιπόν, πολύ που ήσασταν το πρώτο θύμα της ε, ε, παρέμβασής μου, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε. Σας ευχαριστώ πολύ που άμεσα και αμέσως ήρθατε εδώ να μας μιλήσετε εδώ στην Επιτροπή των Προπολογισμών διότι η κατάσταση είναι ανησυχητική. Και δυστυχώς όλες οι πληροφορίες που λαμβάνουμε κατατείνουν στο ότι θα αυξηθούν οι ροές των μεταναστών. Δεν ξέρω πόσο καιρό αντέχει η τρέχουσα πολιτική μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε στο ίδιο μικροσχήματος, μιλούμε την ίδια γλώσσα οπότε και έχουμε συνέστηση των διαστάσεων της κρίσεως. Όμως, αυτό που χρειάζεται είναι μια σφαιρική, πλήρης, ολοκληρωμένη στρατηγική. Χρειαζόμαστε επίσης μια εφόλες της ύλη αναθεώρηση του της εκτίμησης του τοπίου, του σκηνικού σε Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική κλπ. Μια στρατηγική και αυτό θα πρέπει να γίνει τώρα. στην ε, ακρόαση που αφορούσε την ε, Frontex, τι αναφέρθηκε. Ότι χρειάζεται μια πιο μακρόπνοη στρατηγική στα πλαίσια του Horizon 2020 και ότι τούτο θα αργήσει, θα μεταδίθει για το μέλλον. Πάει για το 2020. Οπότε θα πρέπει όμως εμείς από τώρα να αρχίσουμε να δουλεύουμε γιατί είναι και θέμα προϋπολογισμού για των σχετικών κονδυλίων. Όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν σήμερα, ε, τους πόρους για την Τουρκία, για τις χώρες προέλευσης, όλα αυτά απαιτούν ευρηματικές λύσεις. Αλλιώς θα λάβουμε ράπισμα ακόμα χειρότερα από αυτά τα προβλήματα. Επομένως χρειαζόμαστε μια μακρόπνοη, πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και στατική και να ευχαριστήσω την κυρία Γεωργέβα και πάλι. Να τη συγχαρώ επίσης. Νομίζω ότι θα πρέπει να δείξουν υπευθυνότητα τα θεσμικά όργανα και θα πρέπει να ανέβουν μέσω τριμμένου διαλόγου κάποια λύση. Δύο ενστάσει μικρέ. Πρώτα-πρώτα ε, και εγώ να σα ευχηθώ καλώ ορίσατε. Μπράβο που ενεργήσατε ταχύως. Και στη σημερινή κατάσταση απαιτείται να αποδείξουμε στους Ευρωπαίους το ότι ο προπολογισμό θα συμβάλλει στην λύση. Η πρόκληση είναι τεραστία και βέβαια μόνος ο προπολογισμό δεν μπορεί να το λύσει το πρόβλημα. Αλλά είναι ξεκάθαρο το προς προ του Ευρωπαίου ότι ο προπολογισμό θα βοηθήσει κατά δεύτερο λόγο. Να τονίσω αυτό που είπε και ο κύριος Ράινερ Μπέγγι ότι εάν θέλουμε να μην έρθουν και άλλοι πρόσφυγες στους επόμενους μήνες στην Ευρώπη, ε, πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση της χώρας προέλευσης. Είναι ο μόνος τρόπος ούτως ώστε να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή τη συνεχή κρίση. Να σταματήσει ο κόσμος να έρχεται στην Ευρώπη. Θα πρέπει να αυξήσουμε τους πόρους προς αυτές τις χώρες και να βελτιώσουμε τον έλεγχο των δημοσιονομικών της Ευρώπης, να μην υπάρχουν απάτες, και τελικά τα χρήματα να πηγαίνουν σε αυτούς που τα χρειάζονται. Τρεις ερωτήσεις ήθελα πρώτα, σας βλέπω ε, ανήσυχο, οπότε θα μείνω στη μία ερώτηση, μια που να φύγει η Επίτροπος. Είπαμε ότι έχουμε 120 θέσεις παραπάνω για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Τι θα γίνει. Είπαμε για σχέδιο διορθικού προβλησμού για φέτος αλλά συνήθως παίρνει πολλούς μήνες η αύξηση του προσωπικού. Πότε θα μπορέσουν αυτές οι υπηρεσίες να αυξήσουν τους υπαλλήλους τους οι προεπίτροπες. Ευχαριστώ για όλα όσα είπατε. Ας αρχίσουμε από αυτό το τόσο σημαντικό το οποίο είπατε. Δηλαδή, τι μέσα έχουμε να δημιουργήσουμε την κρίση. Δεν ξέρω αυτό είναι καλά για καμαντάτα. Αλλά δεν πρόκειται μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλος ο κόσμος βρίσκεται σε αδυναμία ούτως ώστε να αντιμετωπίσει μια κρίση πολλαπλή. Όταν ε, ε, ε χτύπησε την Τουρκία αυτή η κρίση, τους πρώτους 6 μήνες είχαν 32.000 πρόσφυγες. Και τότε, τότε, τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Γιατί κατασκεύασαν στρατόπεδα που ήταν μια χαρά. Οπότε ε, λέγαμε ότι μπορούμε να φιλοξενήσουμε 50.000 και λέγαμε, μα τι θα γίνει αν μπουν 100.000. Λέγανε, όχι, αποκλείεται. Πού να βρεθούν 100.000 πρόσφυγες. Τώρα όμως έχουμε κοντά στα 2 εκατομμύρια στην Τουρκία. Ίσως ακόμα παραπάνω. Είναι τα επίσημα στοιχεία. 1,9 εκατομμύρια λένε. Τώρα, έξε μια ματιά τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Ε, πάμε από τη μια κρίση στην άλλη. Άρα, Βέβαια, να μην είναι παρηγοριά για μας ότι έχουν και άλλοι κρίσεις να αντιμετωπίζουν. Όμως θα πρέπει και εμείς να προλαμβάνουμε, να προβλέπουμε και να είμαστε πιο ευέλικτοι. Γιατί πρόκειται να χτυπηθεί όλος ο κόσμος από την το του κλίματος και επίσης ε, θα έχουμε και προβλήματα και με τους εξτρεμιστάς. Ακριβώς επί τη βάση των γίνονται σήμερα. Επίσης να δούμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή το πόσο γενναιόδοροι τώρα είναι όλοι. Εγώ είχα προεδρεύσει σε κάποιο όργανο για ανθρωπιστική βοήθεια και παρά το ότι ξέρω τα θέματα, σοκαρίστηκα το ότι το 2000 διατέθηκαν 2 εκατομμύρια δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια και πέρσι 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι ένα άλμα. Οπότε από τα 2,2% ε, του συνόλου του παγκοσμίας της ε, αναψυχής βίδιας πήγε στο 18% πολύ σημαντική αυτή η αύξηση. Ουδέποτε στο παρελθόν είχαμε τέτοια όμως, τέτοια απόσταση, τέτοιο χάσμα μεταξύ αναγκών και χρηματοδότησης. Άρα τι πάνε να πει αυτό. Ότι πρέπει να προχωρήσουμε όσον αφορά την ενίσχυση και να δούμε τι θα κάνουμε με ε, την πολιτική πτυχή του προβλήματος. Και ο καλύτερος τρόπος είναι το να μην γεννάται ανθρωπιστικό πρόβλημα. Το να σβήνουν οι φλόγες του πολέμου. Βλέπω τώρα υπάρχει περισσότερες σοβαρότητα στην αντιμετώπιση. τελευταίες ημέρε να είδαμε τι, τι, τι είπαν και στην Νέα Υόρκη. Το πιο σημαντικό που μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Να ενθαρρύνει. Να προσέχουμε περισσότερο το πώς θα προλάβουμε. Και να ανεσδούμε την δύσκολο οδό της ειρήνευσης. Αυτό το βλέπαμε να έρχεται όμως. Και έγραψε πριν από δύο χρόνια, έφτιαξα ένα blog που έλεγα για τα ταξίδια σε προβληματικές για Λίβανο και Τουρκία και έλεγα για αυτό το κύμα το οποίο έλεγα αργά γρήγορα πρόκειται να έρθει στην Ευρώπη και ότι αν θέλουμε να το αποφύγουμε θα πρέπει να επενδύσουμε εκεί που είναι ο Κοσμάκης ούτω ώστε ε, να μην είναι ο βίος αβίωτος εκεί. Οπότε να και τώρα, τώρα δεν το λέω για μένα. Αυτό σας το λέω για το σύνολο της ανθρωπιστικής κοινότητας που είναι σαν ένα Καναρινάκη στον Τρακοριχείο που λέει υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα. Όμως εμείς αντιδράσαμε με μεγάλη βαρύτητα και άρα τώρα θα πρέπει να σταθεροποιήσουμε τις προσπαθειές μας και να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Όλος ο κόσμος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για αυτή την πολλαπλή, πολύπλευρη κρίση και άρα χρειάζεται όλοι να δεσμευτούν γι' αυτό. Όσον αφορά τώρα τις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πώς θα παρουσιάσουμε το τι κάνει η Ευρώπη. Είπατε, μα έχουμε όλα αυτά τα αρνητικά στοιχεία που κυκλοφορούν και τι σημαίνουν. Γενική Διεύθυνση για τα Δημοσιονομικά ασχολήθηκε με αυτό, να δούμε τι κάνουμε εμείς, τι κάνουν τα κράτη-μέλη, να τα συγκρίνουμε, να τα παρουσιάσουμε και να δείξουμε τι κάνει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να προβάλλεται το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνει πολλά, γιατί άλλοι κάνουν λιγότερο από όσα θα έπρεπε. Ας μην το σχολιάσω. το δεύτερο ερώτημα αφορούσε τα ανεξόφλητα, αν ισχύει το πρόβλημα ναι, ναι, νομίζω ότι ισχύει η ρύθμιση και παρακολουθούμε με προσοχή τις εξελίξεις. Αλλά η τελευταία ανάλυση της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικά έλεγε ότι θα υπάρξουν κάποιες μικρές αλλαγές, αλλά όχι τίποτα το σημαντικό. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να ενημερώνουμε σας Τώρα για την αφιόρωση του πολιτούς πλαισίου δεν μπορώ να σας πω τώρα το χρονοδιάγραμμα για πολλούς λόγους. Να δούμε τι θα κάνουμε την κρίση πρώτα. Να δούμε για τι στρατηγική θα δεσμευτούμε. Μην ξεχνάμε και το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και άλλες μεταβλητές πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ε, επίσης, άλλο ερώτημα αφορούσε τις επιπτώσεις για την αλία. Επρόκειτο για κάποια χρήματα του αποθεματικού. νομίζω 18 εκατομμύρια. Δεν θα υπάρχει συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους, άρα φέτος δεν θα χρειαστούν χρήματα, δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις. Για αυτή τη μείωση 2,2% για την ασφάλεια δεν έχουμε κάποια μείωση. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την υγεία ζώων και φυτών. Δεν καταλαβαίνω. Α, ναι, ε, ε, είχε να κάνει με την ιδιότητα Ευρωπαίου πολίτη, αλλά όχι την ασφάλεια. Πάει η ασφάλεια. Οπότε, τέλος πάντων, νομίζω ότι τα απάντησα όλα και σας ευχαριστώ. Ήταν εξολογη αυτή η ευκαιρία να τα πούμε και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Δεν απάντησα όμως την ερώτηση για τους ελέγχους. Θα πρέπει να αποκτήσουμε περισσότερα μέσα για να υπάρχουν εγγυήσει αξιοποίησης των πόρων και όχι αυτό που κάναμε μέχρι σήμερα. Ναι, θα πρέπει να αναφερθούν οι δημοσιομικοί κανονισμοί. Γιατί ε, έχουν γίνει τόσο δύσκολοι που δεν θέλει κανείς να τους χρησιμοποιήσει και να συνεργαστεί. Για να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο αποδίδει. Και αυτό είναι από τη βάση, bottom up. Οι πολίτε, η διαφάνεια, όλα να είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά, να το μπορεί να τα τσεκάρει οποιοδήποτε και οι νέες τεχνολογίες να χρησιμοποιούμε διαφορετικά. Όχι με αλλεπάλληλους ελέγχους όπως κάνουμε σήμερα και ελέγχους των ελέγχων. γιατί αρχίζει κάτι το 2015 και ολοκληρώνεται ο έλεγχος το 2017 που είναι πια πολύ αργά γιατί έχει, το πράγμα δεν τρέχει πια. Ευχαριστώ και πάλι. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε. Καταλάβαμε ότι όταν ε, ξεσπάει πυρκαγιά δεν θα συζητάμε την τιμή του νερού. Το φόρουμ ε, που έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω ότι έδωσε έμφαση στην βούληση και την προεφημία σας να έχουμε έναν προεπολισμό βάσει αποτελεσμάτων. Εμείς τώρα ε, περιμένουμε να στερέψει, αν θέλετε, να στερέψουν αυτές οι μεταναστευτικές ροές ε, και δεν πρέπει να δούμε μόνο τις επιπτώσεις αλλά και τα αίτια. Και πέρα από τα ε, δημοσιονομικά πέρα από τον προπολισμό υπάρχουν και θεσμικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν. Είπατε να βοηθήσουμε τις αφρικανικές χώρες. Η επιστροφή όμως των ε, τόπων έχει να κάνει με το κατά πόσο θα τους δεχτούν πίσω και στις χώρες τους. Άρα ναι μεν βοήθεια αλλά θα πρέπει ε, και οι δικαιούχοι χώρες αυτών των κονδυλίων να δέχονται τον επαναπατρισμό αυτών των ανθρώπων. Κύριε Γεωργίβα, σας ευχαριστούμε ξανά ε, που ήρθατε σήμερα και έχουμε νομίζω εξαιρετικά επιχειρήματα για την ε, ενδιάμεση αναθεώρηση. Όπως και να χαίρομαι που ο πρόεδρος της Κομισιόν έχει εμπιστευτεί σε μια επίτροπο, τέως επίτροπο αρμόδια για τα ανθρωπιστικά, τα δημοσιονομικά. Τα είχε προβλέψει όλο, ο Ζήτη.